Ε, σας αναφέρω την, την περίπτωση δύο Σουηδών δημοσιογράφων, Πέρσον και Σίμπιερ, που ευτυχώς ε, έφτασαν ε, με ασφάλεια στη Σουηδία. Νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε όλη την χαρά μας για τις αίσθησες εξελίξεις προς τους δύο Σουηδούς δημοσιογράφους. Η κυρία Κορτάτσα Μπίλτ, έχετε να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το λαό της ε, Σουηδίας γιατί απελευθερώθηκαν ο Γιώργο και ο Μάρτιν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ελεγγύη που έδειξαν και την υποστήριξή τους. Ε, τους δόθηκε αμνηστία μαζί με άλλους από τις φυλακές της Αιθιοπίας και επέστρεψαν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Ελπίζω να απελευθερωθούν και όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που κρατούν τις φυλακές ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ενημέρωσαν οι αρμόδιες τσεχικές αρχές ε, για την εκλογή του κυρίου Βόιτσεκ Βίλερ που θα, που θα αντικαταστήσει τον κύριο Γίζη Χάβελ, τον αποβιώσαντα, από την 9η Ιουλίου. Με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2 θα γίνει η... Ε, ε, ο έλεγχος των ασυλιών